Frau Direktorin der η συνεδρίαση. Έχουμε ένα θέμα το οποίο έχει απομείνει την ειδική έκθεση για το θέμα της Ελλάδας και την παρέμβαση της Κομισιόν στην ελληνική ε, δημοσιονομική χρηματοπιστωτική κρίση. Χαν Τάκουλα είναι ο ε, Τον λόγο έχει πρώτα απ' όλα κύριος Μουγκουρούσα. Ε, αγαπητή κυρία Πρόεδρε, αγαπητά μέλη της Επιτροπής Ελέγχου Προϋπολογισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Θα ήθελα να ευχαριστήσω την Επιτροπή σας για την πρόσκληση να σας παρουσιάσω την ειδική έκθεση του Ελεκτικού Συνεδρίου με θέμα την παρέμβαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην ελληνική χρηματοπιστωτική κρίση. Χαίρομαι ιδιαίτερος που θα έχουμε την ευκαιρία να συζητήσουμε μετά την παρουσίαση των πορισμάτων του, ε, του έργου μας. Μάλιστα, η έκθεση αυτή συνιστά τμήμα μια δέσμη ε, ελέγχων που διενεργεί το Ελεκτικό Συνέδριο στα θέματα οικονομική και δημοσιονομική διακυβέρνηση. Μάλιστα, πέρυσι δημοσιεύσαμε μια έκθεση για τη διαχείριση εκ μέρου τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή των Προγραμμάτων Χρηματοδοτική ε, Συνδρομή για την Ιρλανδία, Πορτογαλία, Λετωνία, Ουγγαρία και Ρουμανία. Και μια έκθεση για την τεχνική αρρωγή που χορηγήθηκε στην Ελλάδα με συντονισμό τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Τα προγράμματα που εφαρμόζονται εδώ και 8 περίπου χρόνια στην Ελλάδα, στόχο έχουν την παγίωση μιας υγιούς και βιώσιμης οικονομικής και χρηματοπιστωτικής κατάστασης και την αποκατάσταση της ικανότητας της χώρας να χρηματοδοτηθεί πλήρως στις χρηματοπιστωτικές αγορές. Στον έλεγχό μας εξετάσαμε κατά πόσο η διαχείριση εκ μέρους Ευρωπαϊκής Επιτροπής ε, των προγραμμάτων αυτών ήταν η ενδεδειγμένη και συγκεκριμένα εξετάσαμε διέθετε η Επιτροπή τις κατάλληλες ρυθμίσεις για τη διαχείριση των προγραμμάτων. Σχεδιάστηκαν κατάλληλα και εφαρμόστηκαν αποτελεσματικά οι όροι των τομεακών πολιτικών και εκπλήρωσαν τα προγράμματα προσαρμογής τους κύριους στόχους τους. Ως προς το ενεξελίξη πρόγραμμα, επικεντρωθήκαμε μόνο στα ζητήματα σχεδιασμού. Στο σημείο αυτό θα ήθελα να επισημάνω το εξή. Δεν ελέγξαμε, δεν εξετάσαμε τις ε, πράξεις του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου, ούτε του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Σταθερότητας, ούτε ελέγξαμε τις ενέργειες των ελληνικών αρχών. Σε ό,τι αφορά τώρα την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, επιχειρήσαμε να εξετάσουμε τη συμμετοχή της ΕΚΤ ε, στα ελληνικά προγράμματα οικονομικής προσαρμογής αλλά η τεκμηρίωση που λάβαμε από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα ήταν ανεπαρκής και με τις πληροφορίες αυτές δεν μπορέσαμε να διενεργήσουμε τον έλεγχό μας, μια και το, η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα αφισβήτησε την εντολή του συνεδρίου ως προς το ζήτημα αυτό. Ως εκ τούτου δεν είμαστε σε θέση να αναφερθούμε στο ρόλο της ΕΚΤ στα ελληνικά προγράμματα. Αξιότιμοι Ευρωβουλευτέ. Θα ήθελα να επιστήσω την προσοχή σας στο πρώτο τμήμα της έκθεσης, όπου παρουσιάζουμε τις παρατηρήσεις μας για τον τρόπο με τον οποίο η Ευρωπαϊκή Επιτροπή χειρίστηκε τα προγράμματα. Παρατηρούμε για παράδειγμα ότι κάποιες παραδοχές στα μακροοικονομικά μοντέλα στερούνταν αιτιολόγησης. Σε άλλο παράδειγμα παρατηρήσαμε ότι η τεκμηρίωση για την παρακολούθηση των επισκέψεων ήταν καλή. Θα θέλαμε να είχαμε μπορέσει να διενεργήσουμε παρόμοιες αναλύσεις και για την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα. Παρ' όλα αυτά δεν μας το επέτρεψε η ΕΚΤ. Θα ήθελα να σας υπενθυμίσω ότι αντιμετωπίσαμε παρόμοια κατάσταση στην έκθεση που δημοσιεύσαμε πέρυσι για τον ενιαίο εποπτικό μηχανισμό. Και εκεί η τράπεζα μας παρήχε ελάχιστες πληροφορίες σε σχέση με αυτές που είχαμε ζητήσει για τη διενέργεια του ελέγχου μας. Θα σας κάνω τώρα μια σύντομη επισκόπηση των βασικών απορισμάτων και συμπερασμάτων της έκθεσής μας. Ε, στην αρχή, ο σχεδιασμός του πρώτου προγράμματος έγινε κατεπηγόντος και η διαχείριση και των τριών προγραμμάτων επηρεάστηκε από πολιτικές και οικονομικές αβεβαιότητες. Χρειάστηκε περίπου ένα χρόνο για την Ευρωπαϊκή Επιτροπή προκειμένου να θεσπίσει διαδικασίες. Αρχικά κάποιοι όροι ήταν ασαφείς. Ε, αναγνωρίζουμε όμως ότι με την πάροδο του χρόνου βελτιώθηκε ο σχεδιασμός. Διαπιστώσαμε επίσης ότι οι όροι δεν εντάχθηκαν σε μια ευρύτερη αναπτυξιακή στρατηγική για την Ελλάδα που θα διαρκούσε και μετά τη λήξη των προγραμμάτων. Σε ό,τι αφορά τις μακροοικονομικές παραδοχές, θεωρούμε ότι εσωτερικά ήταν ε, συνεκτικές και ενημερωμένες, αλλά ανεπαρκώς αιτιολογημένες και χωρίς επισημοποιημένες ρυθμίσεις ελέγχου ποιότητας. Μάλιστα, οι προβολές που έγιναν υποτίμησαν εμφανώς την οικονομική κρίση στην Ελλάδα, παρόλο που δεν ήταν μόνη η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αυτή που έπεσε έξω και άλλες ε, διεθνείς οργανώσεις ε, έκαναν παρόμοιες λάθος προβολές. Θα πρέπει να τονιθεί ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή απέδειξε μια πάγια βάση για την ε, παρακολούθηση της εφαρμογής των μέτρων από τις ελληνικές αρχές. Επίσης, ήταν αποτελεσματική συνεργασία με τους λοιπού εταίρου παρά τις περίπλοκες θεσμικέ ρυθμίσει που δεν ε, επισημοποιήθηκαν ουδέποτε προκειμένου να εξασφαλίσουν την απαραίτητη διαφάνεια για το ρόλο και τι ευθύνε των εταίρων. Όπως γνωρίζετε, τα προγράμματα περίχαν κάποιες ε, διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις σε ένα ευρύ φάσμα πολιτικών που κάλυπταν σχεδόν όλες τις λειτουργίες του ελληνικού κράτους. Κατά την αξιολόγηση του σχεδιασμού και της εφαρμογής τέτοιων μεταρρυθμίσεων, επικεντρωθήκαμε σε τέσσερις κέρυες πολιτικές. Τη φορολογία, τη δημόσια διοίκηση, την αγορά εργασίας και τον χρηματοπιστωτικό κλάδο. Στο δεύτερο τμήμα της έκθεσης θα βρείτε μια σειρά παρατηρήσεων για τις ε, ανωτομιακές πολιτικές. Και στην τελευταία τμήμα της έκθεσης επικεντρωνόμαστε στους ιδιαίτερους στόχους των προγραμμάτων και διαπιστώσαμε ότι μόνο σε περιορισμένο βαθμό ε, υλοποιήθηκαν οι στόχοι, εν μέρη λόγω της πολιτικής και οικονομικής αστάθειας ε, της χώρας κατά την περίοδο αυτή. Πρώτα και πάνω απ' όλα, τα προγράμματα αυτά προώθησαν μεταρρυθμίσεις και απέτρεψαν τη χρεοκοπία της χώρας. Αλλά η ικανότητα της Ελλάδας να χρηματοδοτηθεί πλήρως στις χρηματοπιστωτικές αγορές δεν αποκαταστάθηκε. Τα προγράμματα επέφεραν αρκετή δημοσιονομική εξυγίαση και εξασφάλισαν βραχυπρόθεσμη χρηματοπιστωτική σταθερότητα. Μάλιστα, ο χρηματοπιστωτικός κλάδος ε, διαρθρώθηκε, αναδιαρθρώθηκε σημαντικά, αλλά με μεγάλο κόστος. Και τι συστήνουμε σε τελική ανάλυση. Η έκθεσή μας επισημαίνει μια δέσμη 11 συστάσεων που στόχο έχουν να βελτιώσουν την διαχείριση εκ μέρους της Ευρωπαϊκής Επιτροπής οποιοδήποτε μελλοντικού προγράμματος ε, συνδρομής. Ιδιαίτερα συστήνουμε στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή να βελτιώσει τη γενική διαδικασία για το σχεδιασμό των προγραμμάτων συμπεριλαμβανομένης και της διευκρίνησης του ρόλου των εταίρων. Θα πρέπει να ιεραρχήσει πιο αποτελεσματικά τους όρους και να εξασφαλίσει συμπερίληψη των όρων αυτών σε μια ευρύτερη στρατηγική για τη χώρα. Ενώ θα πρέπει ταυτόχρονα να λάβει υπόψη την την, την ε, διοικητική ικανότητα του ενδιαφερόμενου κράτους μέλους. Επίσης, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα πρέπει να αντιμετωπίσει πιο διεξοδικά κάποια κενά δεδομένων και να τεκμηριώσει καλύτερα τις παραδοχές και τις τροποποίησεις των οικονομικών της υπολογισμών. Θεωρούμε ότι τα προγράμματα θα πρέπει να υπόκεινται σε μία αξιολόγηση τουλάχιστον μετά τη λήξη τους. Και εν τέλει συστήνουμε στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή να αναλύσει την κατάλληλη υποστήριξη και το κατάλληλο πλαίσιο εποπτείας για την περίοδο μετά τη λήξη του προγράμματος, λαμβάνοντα υπόψη τι χρηματοδοτικέ ανάγκες της χώρας. Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω θερμά για την προσοχή σας και να σας διαβεβαιώσω ότι είμαι στη διάθεσή σας για οποιασδήποτε απορίες. Σας ευχαριστώ. Σα ευχαριστώ. Είχα δει την έκθεση μετά την δημοσίευσή της. Λοιπόν, υπάρχουν φαντάζομαι πολλές ερωτήσεις. Ο εισηγητής μας είναι ο κύριος ε, Τάκουλα. Έχετε τον λόγο. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Θα ήθελα να ευχαριστήσω το ελεγκτικό συνέδριο για την έκθεση αυτή που βεβαίως χρειάζεται να την συζητήσουμε εις ε, βάθος να έχουμε μια συνολική εικόνα της ε, κατάστασης. Ίσως δεν χρειάζεται να επισημάνουμε ότι η έκθεση αυτή εστιάζει στα, σε μια μεγάλη σε ένα μεγάλο παράγοντα της ε, κατάστασης και βέβαια καλύπτει τις περισσότερες πτυχές της ε, κρίσης. Έχουμε λοιπόν το πρόγραμμα το οποίο κάλυπταν και συντόνισαν Κομισιόν Δέλτα Εντάφη και Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα. Η Κομισιόν λοιπόν ήταν ένας από τους διαχειριστές του προγράμματος ε, χρηματοδότησης. Η έκθεση αναφέρεται σε αυτήν την τρόικα που διαχειρίζεται το πρόγραμμα λέγοντας πως ε, έχει το ελεγκτικό συνέδριο αρμοδιότητα να ελέγξει μόνο ένα από τα θεσμικά όργανα, γι' αυτό ακριβώς και η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα δεν έδωσε τα απαραίτητα παραστατικά. Θεωρώ πως το ζήτημα αυτό της αρμοδιότητας είναι μια άλλη συζήτηση που πρέπει να επιληθεί για καταστάσεις όπως αυτή. Είναι ατυχές γεγονός ότι το Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο δεν έχει πλήρη εικόνα των γεγονότων και ίσως μπορεί να μας ξεκαθαρίσει τα πράγματα. Ένα άλλο θέμα που θίγει η κατάσταση είναι η πολιτική κατάσταση στην Ελλάδα κατά την στιγμή των χρηματοδοτικών προγραμμάτων. αυτή είναι μια λεπτομέρεια την οποία δεν μπορούμε να παραβλέψουμε καθώς αφορά την εφαρμογή των προγραμμάτων που σχετίζεται με τις μεταρρυθμίσεις σε διάφορους τομείς. Νομίζω το σημείο 1 στην έκθεση όπου αναφέρει το ελεγκτικό συνέδριο το επιτόκιο των ελληνικών ομολόγων παράλληλα με τα πολιτικά γεγονότα αντικατοπτρίζει το χάλι στο οποίο βρισκόταν η Ελλάδα. Ελπίζω τώρα να υπάρχει μια ελπίδα για μια πιο θετική κατεύθυνση. Αυτό το οποίο θα ήθελα να ακούσω από το ελεγκτικό συνέδριο είναι ε, που οφείλεται ο χρονισμός της έκθεσης. Μπορεί δηλαδή να μας αιτιολογήσει τον ε, χρόνο και κυρίως την καθυστέρηση στην σύνταξη αυτής της έκθεσης. Ε, η έκθεση συνετάχθη στη μέση της διαδικασίας καθώς ε, το τρίτο πρόγραμμα ακόμα συνεχίζεται και επίσης χρειάστηκαν τρία χρόνια που βεβαίω είναι ένα διάστημα στο οποίο πολλά μπορούν να συμβούν. Για το τρέχον πρόγραμμα τώρα πώς ε, έχουν τα πράγματα. Έχουμε τα ίδια προβλήματα ή αντιμετωπίζουμε άλλα. Κάτι το οποίο θα ήθελα να ακούσω σε αυτή τη συζήτηση είναι και κάποιον από την ελληνική πλευρά. Καλό θα ήταν να υπάρχει και κάποιος από την ελληνική πλευρά που θα σχολιάσει το ζήτημα. Θεωρώ ότι ε, το η συνεισφορά της ελληνικής πλευράς ε, στην ε, επιτυχία των μεταρρυθμίσεων είναι ζωτικής σημασίας. Ε, πρέπει λοιπόν προγράμματα όπως αυτό εδώ να τα διαχειριζόμαστε με τρόπο διαφανή. Βεβαίως ελπίζουμε ότι αυτό είναι το τελευταίο, αλλά εάν υπάρξει ανάγκη για άλλο πρόγραμμα στο μέλλον, νομίζω ότι η διαφάνεια είναι ένας παράγον κλειδί. Αυτά από εμένα. Yeah. Σας ευχαριστώ. Σημαντικά ερωτήματα νομίζω, τα οποία θα μπορούσε να απαντήσει αμέσως η Κομισιόν και μετά το ελεγκτικό συνέδριο και μετά ε, έχουν ζητήσει τον λόγο 8 συνάδελφοι. Παρακαλώ. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε που μου δίνετε το λόγο. Κυρία Πρόεδρε, αγαπητά μέλη της Επιτροπής, η Κομισιόν Δεύτερος ορίζει αυτή την ειδική έκθεση του ελεγκτικού συνεδρίου που όπως μας υπενθύμεσε το μέλος του ελεγκτικού συνεδρίου καλύπτει τον σχεδιασμό και την εφαρμογή των δύο πρώτων προγραμμάτων στήριξης αλλά μόνο τον σχεδιασμό του τρέχοντος προγράμματος. Ο συνήθως η Κομισιόν βεβαίω δέχεται την επικοδομητική ανάλυση των δραστηριοτήτων της και δέχεται συστάσεις για το πώς μπορούν να υπάρξουν βελτιώσεις στον σχεδιασμό προγραμμάτων οικονομικής στήριξης. Και για τον λόγο αυτό η Κουψιόν δέχεται όλες τις συστάσεις του ελεγκτικού συνεδρίου και θα τις εφαρμόσει μέχρι το τέλος του 2018. Ε, ενώ βεβαίω πολλές ε, από αυτές τις συστάσεις εφαρμόζονται ήδη στο υφιστάμενο πρόγραμμα του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού ε, Σταθερότητας και ήδη η Κομισιόν όπως βλέπετε και στις απαντήσεις μας είχε ήδη αντιδράσει σε αυτές τις συστάσεις. Και αυτή είναι μια πρώτη απάντηση στις ερωτήσεις του εισηγητή. Τώρα, θα ήθελα να δώσω δύο παραδείγματα για να σας ε, δείξω το πώς εφαρμόζουμε δύο συστάσεις. Πρώτα απ' όλα το παράδειγμα της σύστασης υπαριθμών 2 που λέει ότι η Κομισιόν θα πρέπει να οργανώσει καλύτερα τις προτεραιότητες για τα συγκεκριμένα μέτρα τα οποία αφορούν την ισορροπία εκείνη για την επίτευξη των στόχων των προγραμμάτων. Να υπενθυμίσω ότι πριν δεσμευτούν σε οποιοδήποτε όρους οι ελληνικές κυβερνήσεις και υπογράψουν ένα μνημόνιο συναντήληψης, ε, όλοι οι όροι συζητούνται και συμφωνούνται με τις αρχές ε, και στο τεχνικό και στο πολιτικό επίπεδο για να διασφαλιστεί μια σαφής και κοινή αντίληψη και βεβαίως ε, πάρα πολύ σημαντικό αυτό να υπάρχει και μια προσήλωση στην διαδικασία των μεταρρυθμίσεων. Ενώ λοιπόν κάποιοι όροι γενικά εκφράζονται γενικόλογα και υπάρχουν σαφείς τελικοί στόχοι, κατόπιν συντάσσονται πιο συγκεκριμένες κατευθυντήριες γραμμές που περιγράφουν τα μέσα και τα βήματα εφαρμογής αυτών των μεταρρυθμίσεων. Τώρα, αυτή τη στιγμή στο πρόγραμμα του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Σταθερότητας έχει εισαχθεί η έννοια των παραδοτέων κλειδιών, όπως λέγονται, για να υπάρχουν σαφείς κατευθυντήριες γραμμές για το ποια μέτρα απαιτούνται επιγόντως και είναι πρώτης προτεραιότητας. Οπότε βλέπετε ότι είμαστε ήδη σε μια διαδικασία ενσωμάτωση αυτών των μαθημάτων. Δεύτερο παράδειγμα, εάν μου επιτρέπετε, για τη σύσταση παριθμών 8 που λέει η Κομισιόν θα πρέπει να είναι πιο συστηματική στην αξιολόγηση της ικανότητας της διοίκησης ε, των κρατών μελών για να εφαρμόσουν τις μεταρρυθμίσεις και στην ανάγκη για τεχνική αρρωγή. Ε, εδώ πέρα να πω ότι δεν έχουμε μόνο αξιολογήσει την ικανότητα αυτή, αλλά βοηθούμε και έχουν γίνει σοβαρές προσπάθειες ε, ευθύς εξ αρχής για να αντιμετωπιστούν οι ελλείψεις στην διοικητική ικανότητα, παραδείγματο χάνει με τη σύσταση της Task Force για την Ελλάδα. Επίσης, έχει υπάρξει τεχνική υποστήριξη σύμφωνα με, τις, ε, με τους όρους του τρέχοντος προγράμματος, όπου έχουμε την στήριξη σε διάφορες μεταρρυθμίσεις και η βοήθεια αυτή έχει περιληφθεί ρητός στο μνημόνιο αυτό συναντήληψης. Και μέσα σε τρεις μήνες από την ε, οριστικοποίηση του προγράμματος, η Κομισιόν συμφώνησε με τις ελληνικές αρχές ένα σχέδιο τεχνικής συνεργασίας για να υποστηριχθούν αυτές οι διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις. Η υπηρεσία υποστήριξης των διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων εντός της Κομισιόν που είναι 190 άτομα, είναι μια ολόκληρη υπηρεσία, παρέχει υποστήριξη στα κράτη-μέλη και συγκεκριμένα στις ελληνικές αρχές σχεδόν σε όλους τους τομείς που περιέχονται στο πρόγραμμα. Οπότε βλέπετε πως έχουμε κάνει πολλά από την πλευρά της βοήθειας. Όπως είπε τώρα και το μέλος του Ελεκτικού Συνεδρίου, να υπενθυμίσω τους στόχους του προγράμματος ε, βοήθειας. Στόχο έχει να δημιουργήσει χρηματοπιστωτική σταθερότητα και να αποκαταστήσει την πρόσβαση στις αγορές. Εκφύσεως λοιπόν τα προγράμματα αυτά δημιουργούνται σε στιγμές οξίας κρίσης όπως έγινε και στην Ελλάδα. Αλλά έχει μεγάλη σημασία να λαμβάνουμε υπόψη την οικονομική και την πολιτική κατάσταση και πλαίσιο του κάθε προγράμματος εντός του οποίου έγιναν οι συγκεκριμένες επιλογές πολιτικής. Και να θυμόμαστε επίσης ε, το ιστορικό των γεγονότων. Και άρα ως τελικό συμπέρασμα θα ήθελα να αναφερθώ στην εισαγωγική πρόταση του ελεγκτικού συνεδρίου που λέει στο δελτίο τύπου. Τα προγράμματα αυτά συμφωνήθηκαν με την Ελλάδα, έδωσαν πρόθεσμη χρηματοπιστωτική σταθερότητα και κατέστησαν δυνατή κάποια πρόοδο στις μεταρρυθμίσεις. Λοιπόν, θα σταματήσω εδώ και είμαι στη διάθεσή σας για ερωτήσεις. Και Μογκορούτσα, θέλετε κι εσείς να τοποθετηθείτε για αυτά τα οποία ρώτησε ο εισηγητής. Ε, Χωρίς μικρόφωνο, δυστυχώς. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Ο εισηγητής αναφέρθηκε σε πολύ σημαντικά ζητήματα. Να ξεκινήσω με την ημερομηνία δημοσίευσης της έκθεσης. Τη διάρκεια της και να πω ότι δεν ήταν καθόλου εύκολη η εκπόνηση της έκθεσης αυτής. Ο στόχος μας ήταν ένας κινούμενος στόχος. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ήταν απασχολημένη με το δεύτερο πρόγραμμα που έμεινε ανολοκλήρωτο και γι' αυτό το λόγο συμπεριλάβαμε τα ζητήματα σχεδιασμού του τρίτου προγράμματος στην έκθεσή μας. Επίσης, έχουμε δημοσιεύσει και άλλες συναφείς εκθέσεις με την ειδική αυτή έκθεση. Θα θυμάστε την έκθεσή μας για τα προγράμματα της Ιρλανδίας, της Πορτογαλίας, της Ρουμανίας, ε, Λιθουανίας και Ουγγαρίας. Από αυτή την άποψη, η περιπλοκότητα των ελληνικών προγραμμάτων οδήγησε στην καθυστέρηση στην υποβολή της τελευταίας έκθεσης. Εν τω μεταξύ όμως, καταρτήσαμε και άλλες εκθέσεις από τα μαθήματα που αντλήσαμε από την εφαρμογή των ελληνικών προγραμμάτων. Είχαμε για παράδειγμα την έκθεση σε ό,τι αφορά την Task Force για την Ελλάδα, δηλαδή την ε, τεχνική αρρωγή που πρόσφερε στην Ελλάδα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και εκεί είχαμε σημαντικές συστάσεις για το σχεδιασμό των προγραμμάτων ε, τεχνικής αρρώγης για το μέλλον. Θεωρώ ότι η ημερομηνία δημοσίευσης ε, της έκθεσης ε, είναι σωστή. Μια και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δέχτηκε τις συστάσεις μας και θα τις αξιοποιήσει στο σχεδιασμό νέων προγραμμάτων. Θα χρειαστούν λοιπόν για το μέλλον, αλλά ήδη χρησιμοποιούνται οι συστάσεις μας στην διαδικασία παρακολούθησης του τρέχοντος προγράμματος. για την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα. Στην έκθεση εξηγούμε με σαφήνεια ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και άλλα θεσμικά όργανα προβλέπουν την παροχή ε, τεχνικής αρρωγής ε, για ένα πρόγραμμα που καταρχήν ε, ε, εναπόκειται στις ελληνικές αρχές, τις αρχές που το χρηματοδοτούν και αυτές είναι υπεύθυνε με την διεξαγωγή και την εφαρμογή των μεταρρυθμίσεων. Η ανάλυση στην έκθεσή μας περιορίζεται στο έργο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Ε, για τον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Σταθερότητας γνωρίζετε ότι εμείς δεν έχουμε αρμοδιότητα το Ευρωπαϊκό Ελεκτικό Συνέδριο δεν έχει αρμοδιότητα ελέγχου του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Σταθερότητας. Σε ό,τι αφορά την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, έχουμε κάποιες αρμοδιότητες, αλλά είναι περιορισμένες. Οι αρμοδιότητες μας περιορίζονται μόνο στην ε, επιχειρησιακή αποτελεσματικότητα της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας. Παρόλα αυτά, στα πλαίσια αυτών των περιορισμένων αρμοδιοτήτων μας δεν καταφέραμε να διεκπαιρεώσουμε το έργο μας. Και αυτό προβλημάτισε ιδιαιτέρως ε, το ελεγκτικό συνέδριο, γιατί δεν είναι η πρώτη φορά που προσκρούμε σε τέτοια αντίσταση από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα. Στην έκθεση για τον ενιαίο εποπτικό μηχανισμό των τραπεζών, επίσης είχαμε πρόβλημα, κάποιες δυσκολίες. Και μάλιστα στο, Ευρωπαϊκό... Ευρωπαϊκό Ελεκτικό Συνέδριο. Αυτή τη στιγμή ε, μελετούμε διεξοδικά πώς θα πρέπει στο μέλλον να δράσουμε απέναντι στην Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα για να ξεπεράσουμε αυτό το διέξοδο ή ενδεχομένως και εφόσον χρειαστεί να προασπίσουμε τις ελεκτικές μας δραστηριότητες που είναι ένα καθήκον που μας το επιβάλλει η συνθήκη απέναντι στην Ευρωπαϊκή Κοινή Γνώμη απέναντι στους ενδιαφερόμενους και στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Οφείλουμε να γνωμοδοτήσουμε για την επιχειρησιακή αποτελεσματικότητα της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας. Οι ελληνικές αρχές βρίσκονται εκτός του πεδίου ελέγχου του ελεκτικού συνεδρίου. Στην έκθεση πάντως αναγνωρίζουμε ότι η πολιτική αστάθεια επηρέασε αισθητά την υλοποίηση των στόχων του προγράμματος. Και το γεγονός ότι το δεύτερο πρόγραμμα δεν έκλεισε, έμεινε ολοκλήρωτο. οφειλόταν εν μέρη σε δύσκολες πολιτικές συνθήκες και αυτό το αναφέρουμε στην έκθεσή μας. Και από αυτήν την άποψη, όταν εξετάζουμε την εμβέλεια της έκθεσής μας, θα ήθελα να αναγνωρίσω και να σας ευχαριστήσω θερμά τις υπηρεσίες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την πολύ αγαστή συνεργασία που είχαμε. Εμείς εκφέρουμε μια γνώμη προσπαθώντας να εξασφαλίσουμε διαφάνεια και λογοδοσία για περίπλοκα προγράμματα. Είχαμε πρόσβαση σε εσωτερικές διαδικασίες, ε, στους υπολογισμούς της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και μερικές φορές μάλιστα οι υπηρεσίες ε, ε, χρειάστηκε να εργαστούν υποπίεση λόγω των όρων του προγράμματος. Πάντως ε, ήταν πολύ συνεργάσιμη η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και αυτή η ενημέρωση που είχαμε για, την, ε, για τις εσωτερικές διαδικασίες, για την ε, επιχειρησιακή αποτελεσματικότητα της ΕΚΤ και τη συμβολή, του τη συμβολή της στην Ευρωπαϊκή Κεντρική, ε, στην, στο ελληνικό πρόγραμμα, μόνο αυτό το τμήμα έμεινε ε, ατελές, ανολοκλήρωτο. Σε ό,τι φορά τη συνεργασία με τα, τους εταίρους που συμβάλλουν στο πρόγραμμα, επαναλαμβάνουμε τη σύσταση που είχαμε διατυπώσει και σε προηγούμενα προγράμματα. Δηλαδή ότι στο μέλλον καλό θα ήταν να επισημοποιηθεί αυτή η συνεργασία για να γίνει μια σαφής κατανομή των ευθυνών και των ρόλων για να έχουμε μεγαλύτερη διαφάνεια και να διευκολυθεί και η λογοδοσία η συνεργασία με το Διεθνές Ομισματικό Ταμείο, με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και με την Τράπεζα ήταν ουσιαστική και αποτελεσματική και αυτά τα διατυπώσαμε στην έκθεσή μας. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ. Πέντε μέλη της Επιτροπής ε, έχουν ζητήσει το λόγο και τρεις Έλληνες συνάδελφοι που δεν είναι μέλη της Επιτροπής, αλλά βεβαίως τους ενδιαφέρει το θέμα που έχουν ζητήσει να μιλήσουν. Προτείνω λοιπόν δύο λεπτά για τον καθένα και και 30 θα τελειώσει η συνεδρίαση γιατί μετά έχουμε τον τριμερή διάλογο. Λοιπόν, ξεκινάει ο κύριος Σντεχόφσκι. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Ξέρετε ότι πάντα σας σέβομαι, αλλά δύο λεπτά για να πω αυτά τα οποία είχα να πω για αυτή την έκθεση δεν είναι δυνατόν. Τέλος πάντων θα προσπαθήσω. Γνωρίζετε ότι ε, σας ε, σέβομαι. Πρώτα απ' όλα ε, για την Ελλάδα πρέπει να διαπιστώσουμε ότι πρέπει να ληφθεί υπόψη ότι πολλά προγράμματα ε, τα προγράμματα ελαμβάνουν υπόψη βεβαίω το σε ποια χρονική στιγμή ξεκίνησαν. Και βεβαίως υπήρχαν και μακροπρόθεσμα εσωτερικά προβλήματα της ε, Ελλάδος. Μεταξύ 2009 και 2015 έγιναν έξι φορές εκλογές στην χώρα. Οπότε υπήρχε εδώ πέρα μια ολόκληρη παλέτα οικονομικών μέτρων, διαρθρωτικών μέτρων, τα οποία όμως δεν μπόρεσαν να εφαρμοστούν, γιατί με τέτοιες πολιτικές αλλαγές είναι σαφές ότι δεν μπορεί να είναι αποτελεσματική εφαρμογή των προγραμμάτων. Οπότε βλέπουμε μια κακή ε, χαμηλή αποτελεσματικότητα των ε, διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων. Και έτσι καταλήγουμε στο συμπέρασμα ότι υπάρχει κακός συντονισμός ε, όσον αφορά και την ε, εφαρμογή των προγραμμάτων. Επίσης ε, δεν ε, καταλαβαίνω γιατί οι σχέσεις ε, είναι μόνο άτυπες και γιατί δεν έχουμε ξεκάθαρο καθορισμό των αρμοδιοτήτων και ξεκάθαρες διαδικασίες. Μπορεί να μας τα εξηγήσει αυτά η Κομισιόν. Και επίσης μια ερώτηση εξακολουθεί η Ελλάδα να βρίσκεται σε κρίση. Ευχαριστώ. Ε, ναι. Δύο λεπτά είναι εντάξει για δύο ερωτήσεις. Η πρώτη μου ερώτηση αφορά κάτι που συμπεριλαμβάνεται και στην έκθεση, ότι δηλαδή η Κομισιόν πολιτικός καθοδηγήθηκε σε μεγάλο βαθμό από το Eurogroup και από τις αποφάσεις που έλαβε αυτό. Οπότε συμφωνώ με την ερώτηση του εισηγητή προς εσάς και ίσως και προς το ελεγκτικό συνέδριο. Σε ποιο βαθμό μπορούμε να εστιάζουμε μόνο στην Κομισιόν χωρίς να λαμβάνουμε υπόψη ολόκληρη τη διαδικασία που εν μέρη ήταν διαφανής αλλά εν μέρη καθόλου στο σχεδιασμό δηλαδή και στην εφαρμογή αυτών των προγραμμάτων. Θα ήταν ενδιαφέρον να γνωρίζουμε σε ποιο βαθμό ε, με ευχαρίστηση ακολούθησε η Κομισιόν αυτές τις κατευθύνσεις, ε, οι οδηγίες, ε, ας τις από το Eurogroup. Η δεύτερη μου ερώτηση έχει να κάνει με τη μεταρρύθμιση της αγοράς εργασίας. Ένα από τα ζητήματα που ήταν τα πιο επίμαχα ήταν η αποκατάσταση των συλλογικών διαπραγματεύσεων. ακόμα και μετά την κατάληξη που είχε, στην οποία είχε φτάσει ο ειδικό απεσταλμένο ότι οι προτάσει τη ελληνική κυβέρνηση ήταν σύμφωνε με τι αρχικέ προτάσει, υπήρχε μία ε, άρνηση παρατεταμένη για τι συλλογικέ διαπραγματεύσει. Αυτό σημαίνει ένα είδο ε, ε καθήλωση σε οικονομικά και ε, χρηματοπιστωτικά μέτρα υπό τον αιγίδα της λιτότητας που όμως αρνήθηκαν τις σε συλλογικέ διαπραγματεύσεις, πράγμα που θα μπορούσε ίσως να έχει αμβλύνει ε, το κοινωνικό κόστος. Τι γίνεται λοιπόν με αυτό το πολιτικό δόγμα και γιατί δεν αποκαταστάθηκαν οι συλλογικέ διαπραγματεύσεις πολύ νωρίτερα. Ευχαριστώ. Υποδειγματικός. Ο κύριος Μαριάς παρακαλώ. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Θα προσπαθήσω στα δύο λεπτά να τοποθετηθώ σε αυτό το θέμα το οποίο ταλανίζει την Ευρώπη αλλά κυρίως ταλανίζει τον ελληνικό λαό εδώ και 7 χρόνια. Τρία προγράμματα, τρία μνημόνια τα οποία απέτυχαν. Έχουμε αυτή τη στιγμή το 40% του πληθυσμού να ζει κάτω από τα όρια της φτώχειας. Την ανεργία έχει φτάσει στο 26-27%. Οι μισθοί έχουν μειωθεί 40%, το ίδιο και οι συντάξεις ε, έχουν κλείσει χιλιάδες μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Επομένως το πρόγραμμα, όπως λέγεται, τα μνημόνια, η συνταγή του μνημονίου έχει αποτύχει. Και απέτυχε για τον απλό λόγο ότι στόχος δεν ήταν η διάσωση της ελληνικής οικονομίας, αλλά όπως παραδέχθηκε και ο κύριος Ντάισεμπλουμ, ήταν η διάσωση των τραπεζών διότι διασώθηκαν οι ελληνικές και γερμανικές και γαλλικές και υπόλοιπες τράπεζες που είχαν ομόλογα του ελληνικού δημοσίου. Οι ξένες τράπεζες είχαν 150 δισεκατομμύρια ευρώ ομόλογα, διασώθηκαν και φυσικά φτωχοποιήθηκε ο ελληνικός λαός, λαιλατείται η δημόσια περιουσία, διαλύθηκε η οικονομία και κανένας δεν ενδιαφέρεται. Για σας φέρω ένα παράδειγμα, η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα κατάφερε στο PSI να εξαιρέσει τα δικά της ομόλογα, τα οποία ήταν κοντά στα 54 δισεκατομμύρια ευρώ ονομαστική αξία και έτσι γλίτωσε. Και το κούρεμα το υπέστησαν οι μικροομολογιούχοι, το υπέστησαν τα ελληνικά ασφαλιστικά ταμεία κλπ. Και όχι μόνο αυτό, αλλά η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα έχει αγοράσει αυτά τα ομόλογα με έκπτωση 40% και τα πληρώνεται στο 100%. Και αφού τα πληρώνετε αυτά. Η Ελλάδα δεν έχει να πληρώσει αυτά τα ομόλογα. Ξαναπαίρνει νέο δάνειο, νέο μνημόνιο. Αυτό λοιπόν είναι ένα τρίκ όπου οι δανειστέ πλέον έχουν καθυποτάξει τη χώρα. Και το βασικό σε σχέση με την Κομισιόν είναι ότι βρίσκεται σε σύγκρουση συμφερόντων. Διότι έχει αναλάβει να εφαρμόσει ένα μνημόνιο που οι ίδιοι ξέρουν ότι είναι λάθο, οι ίδιοι παραδέχτηκαν ότι έκαναν λάθο στον πολλαπλασιαστή, οι ίδιοι έχουν ομολογήσει ότι έβαλαν λάθο συνταγή, αλλά δεν ενεργούν I'm going to finish in 30 uh, seconds really. Αλλά δεν ομολογούν ότι ενεργούν ως εντολοδόχοι των δανειστών και όχι ως θεσμός ο οποίος υπερασπίζει το κοινοτικό δίκαιο και παραβιάζονται τα δικαιώματα των Ελλήνων πολιτών, παραβιάζονται οι διατάξεις για την προστασία των θεμελιωδών δικαιωμάτων και η Κομισιόν κάνει ότι δεν καταλαβαίνει και ότι δεν ξέρει. Πρέπει λοιπόν, θα τελειώσω, πρέπει λοιπόν αυτή η κομμωδία να σταματήσει και να γίνει αποδεκτό ότι έχει ευθύνε η Ευρωπαϊκή Ένωση και πρέπει να αποζημιώσει τον ελληνικό λαό για αυτή τη ζημιά την τεράστια που έχει υποστεί. Ευχαριστώ. Collega Σας ευχαριστώ. Είναι πολύ σημαντική αυτή η έκθεση. Ακούω ότι θα ακολουθήσει και άλλη μια έκθεση και βεβαίως εδώ πέρα θα πρέπει οι συντονιστές να συνοηθούμε να το συζητήσουμε το θέμα σοβαρά, όχι σε τόσο σύντομο χρονικό διάστημα. Δεν νομίζω ότι είναι σωστό αυτό το οποίο κάνουμε ως ε, Επιτροπή. Το πρωί ήμουν στην ΑΦΚΟ όπου συζητήσαμε έκθεση για τα θεμελιώδη δικαιώματα και έπρεπε να έρθω εδώ γιατί βεβαίως ε, είναι πολύ σημαντική αυτή η έκθεση και δεν αξίζει νομίζω αυτή η πολύ σύντομη παρουσίαση σαν να ήταν ένα σύντομο έγγραφο εργασία. Δεύτερον, κάτι το οποίο επίση είναι πάρα πολύ σημαντικό και πολιτικό, λέει το ελεγκτικό συνέδριο, ναι, εμεί έχουμε αρμοδιότητα να ελέγξουμε την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα ή τουλάχιστον τη λειτουργική αποτελεσματικότητα. Αυτό δεν συνέβη, αρνείται η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα. Εδώ πέρα πρέπει να βοηθήσουμε εμεί ω Κοινοβούλιο το ελεγκτικό συνέδριο. Δεν μπορούμε να αποδεχτούμε ότι η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα αρνείται ε, να ελεγχθεί και η έκθεση τελικά να ελέγχει μόνο την Κομισιόν και όχι τα υπόλοιπα μέλη του προγράμματος. Τώρα όσον αφορά το περιεχόμενο της ε, έκθεσης, ε, οπωσδήποτε θα έχουν να πούν πολλά περισσότερα και Έλληνες συνάδελφοι. Βλέπουμε αυτό το οποίο Έγινε δηλαδή ότι ήρθε η Κομισιόν, έπρεπε να κινηθεί γρήγορα, υπάρχουν διάφορες υπηρεσίες και η κάθε μία κάνει το δικό της. Και το λέει το ελεγκτικό συνέδριο και επίσης δεν έγινε μία ε, ε, αξιολόγηση του κοινωνικού αντικτύπου. Ε, επίσης, ευτυχώς από ό,τι λέει η Κομισιόν έγιναν δεκτές και εφαρμόστηκαν όλες οι συστάσεις, αλλά πρέπει να αφιερώσουμε περισσότερο χρόνο σε αυτό. το. Ευχαριστώ. Κοιτάξτε, πρόκειται για πολύ ε, μακροσχελή παρουσίαση. Κανονικά τις εκθέσεις αυτές κοιτάμε σε 30 λεπτά. Τώρα αφιερώσαμε μια ώρα. Δεν ξέρω εάν δεν επαρκεί, γιατί η ποιότητα των επιχειρημάτων... Τέλος πάντων. Ο κύριος Φλάναγκαν από εμά, η ποιότητα των επιχειρημάτων. Λυπούμε που άκουσα κάτι τέτοιο. Εν πάση περιπτώσει, η πρότασή μου είναι να πάρουμε αυτή την έκθεση και να την πετάξουμε στα σκουπίδια και να ξαναρχίσουμε. Γιατί ρωτάμε πολλά ερωτήματα, αλλά πουθενά εδώ δεν βλέπω καμιά αναφορά στα κονδύλια που πήγαν στο ελληνικό πρόγραμμα. 250 σχεδόν δίση. Και όπω όλοι γνωρίζουμε πάρα πολύ καλά, αυτά τα χρήματα δεν ήταν όλο το ποσό, ήταν κάποιο κομμάτι που χρησιμοποιήθηκε πάρα πολύ αποτελεσματικά από την Ευρωπαϊκή Ένωση για να παρενοχλήσει και να αναγκάσει την ελληνική κυβέρνηση να δεχτεί διαδοχικά προγράμματα που αποδείχθηκαν καταστροφικά για τον ελληνικό όλα, ο πάντοτε υπάρχει λόγος για να μην τα κάνεις όλα αυτά. Ο απλός άνθρωπος ε, δεν μπορεί να προστατευτεί ποτέ. Γιατί λοιπόν να μην κάνουμε μια ιατροδικαστική εξέταση, να δούμε πού πήγαν στην Ιρλανδία. 67,5 δις από την Τρόικα δόθηκαν στην Ιρλανδία. Ένα ε, ποσά τα οποία βάλαμε στις τράπεζές μας ήταν ακριβώς τα ίδια και ξέρουμε τουλάχιστον πού πήγαν τα λεφτά, ποιος ακριβώς γλίτωσε. Οι τράπεζες, όχι μόνο οι Ιρλανδικές, αλλά ολόκληρο του κόσμου οι τράπεζε τράπεζες, οι τράπεζες ειδικά της Ένωσης. Πού πήγαν λοιπόν τα ελληνικά ε, δισεκατομμύρια, πού κατέληξαν, έγινε πρόσφατα μια μελέτη από Γερμανικό Πανεπιστημίο που κατέληξε ότι 90% των τραπεζών και πάνω από το 90%, όχι μόνο ελληνικέ τράπεζε, τράπεζε σε ολόκληρη την Ευρώπη, στη Γερμανία και στη Γαλλία ειδικά, τα πήραν. Και μόνο το 5% των διεθνών χρημάτων ε, που χρησιμοποιήθηκαν για τη διάσωση τη Ελλάδα ε, κατέληξαν στην πραγματική οικονομία τη χώρα. Λιγότερο από 10 εκατοδείς ε, κατέληξαν στα ελληνικό κρατικό ταμείο, ε, λέει αυτή η ίδια μελέτη. Αυτή η έκθεση λοιπόν είναι ένα, ένα ασβέστομα όλης της κατάστασης για να καλυφθούν τα όσα έγιναν τα, αυτή η έκθεση δεν είναι τίποτα παραπάνω και όσοι ήθιστε υπάρχουν πάντοτε κάποιοι τεχνικοί λόγοι γιατί οι απλοί άνθρωποι στην ουσία την πατάνε γιατί είναι πάρα πολύ περίπλοκα όλα αυτά τα πράγματα υποτίθεται. Δύο ακόμα μέλη δεν είναι μέλη κύριος παρακαλώ. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Ε, η ανάγνωση και η ανάλυση της έκθεσης μας δημιούργησε έκπληξη τη στιγμή που όχι μόνο ο κύριος Ντάιζελμπλουμ πρόσφατα δήλωσε ότι αυτά τα προγράμματα διαμορφώθηκαν όχι για αλληλεγγύη και στήριξη της Ελλάδας αλλά για τη λύση των προβλημάτων και τη σωτηρία των Ευρωπαϊκών Τραπεζών και του Ευρώ ήταν και ο κύριος Όλι Ρεν, απευθύνομαι στην εκπρόσωπο της Κομισιόν, που είχε παραδεχτεί το ίδιο πράγμα το 2014. Έρχεται λοιπόν αυτή η έκθεση που κατά μία έννοια εμφανίζει το πρόβλημα υποτίθεται τεχνικό αλλά είναι πολιτικό και θέλει να μας πει δηλαδή και την ευρωπαϊκή και την ελληνική κοινή γνώμη ότι για την αποτυχία των ελληνικών προγραμμάτων για τη συνέχιση του φαύλου κύκλου ύφεση, λιτότητας, ανεργίας ύφεση φταίει ο κακός σχεδιασμός, οι κακές ελληνικές κυβερνήσεις που καθυστερούσαν στις μεταρρυθμίσεις γιατί μετρούσαν το πολιτικό κόστος και δεν φταίει αυτό που είναι κατά τη γνώμη μου φανερό, οι πολιτικέ τη Ευρωπαϊκή Ένωση, οι πολιτικέ του Συμφώνου Σταθερότητα και τη ενία αγορά. Το πρόβλημα λοιπόν είναι πολιτικό. Αναφέρομαι συγκεκριμένα σε δύο πράγματα ακόμα για να δείξω το πώς καταλήγει αυτή η έκθεση σε αυτά τα συμπεράσματα. Λέτε λοιπόν ε, κύριοι του ε, Ελεκτικού Συνεδρίου ότι αυτά τα δύο προγράμματα της Ελλάδας τουλάχιστον τα πρώτα δεν είχαν ενταχθεί σε μια ευρύτερη στρατηγική Τη στιγμή που η συνταγή όμως της Κομισιόν για την ύφεση στην Ευρωπαϊκή Ένωση είναι η ίδια. Τα ίδια ζητάει η Κομισιόν από την Ελλάδα, από τη Γαλλία, περικοπές κρατικών δαπανών, ιδιωτικοποίηση, ελαστικοποίηση εργασιακών σχέσεων, μείωση των μισθών με απότερο σκοπό τις ιδιωτικές επενδύσεις. Δεύτερο, αναφέρεστε ότι το ελληνικό τραπεζικό σύστημα απορρόφησε 45 δις ευρώ για ανακεφαλοποίηση. Την ίδια στιγμή που είναι η ίδια η Ευρωπαϊκή Ένωση που σχεδίασε το καταστροφικό κούρεμα που έπληξε άνισα τις ελληνικές τράπεζες σε σχέση με τις υπόλοιπες ευρωπαϊκές τράπεζες και που πρόλαβαν να πουλήσουν τα ελληνικά ομόλογα της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας πριν το κούρεμα. Επομένως τελειώνω. Την αλήθεια κύριε. Και την οφείλετε την, οφείλετε, την οφείλουμε και στην ελληνική κοινή γνώμη και στην ευρωπαϊκή κοινή γνώμη. Όχι, όχι αυτή αυτής της κατάστασης, η οποία δεν είναι μόνο για την Ελλάδα. Ευχαριστώ πολύ που με ακούσατε. Σας ευχαριστώ. Ναι, κύριος Παπαδημούλης. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Το Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο με την έκθεσή του, που τη θεωρώ μια θετική δουλειά, καταγράφει λάθη στο σχεδιασμό του προγράμματος, αποτυχία παταγώδη στις βασικές του προβλέψεις και διαπιστώνει και ένα έλλειμμα διαφάνειας και δημοκρατικής λογοδοσίας που διαρκεί ακόμη και σήμερα και έρχεται να καταλήξει στο ίδιο συμπέρασμα που ομολόγησε ο κύριος Ντάισεμπλουμ πριν μερικές εβδομάδες δημόσια. Θα προτιμούσα όμως ο κύριος Ντάισεμπλουμ αυτά που μας είπε ότι το κάναμε για τις τράπεζες αυτό να τα έλεγε τότε που είχε δύναμη ως πρόεδρος του Eurogroup και αποφάσιζε και όχι τώρα λίγο πριν τη λήξη της θητείας του. Και τα λάθη αυτά στο σχεδιασμό και την αποτυχία στις προβλέψεις την έχει πληρώσει με βαρύτατο τίμημα κυρία Πρόεδρε και σας παρακαλώ μην υποτιμάτε αυτά τα επιχειρήματα όταν ακούγονται. Ο ελληνικός λαός, το ανθρώπινο και το κοινωνικό τίμημα αυτών των λαθών και αυτής της αποτυχίας των προβλέψεων είναι τεράστιο. Μπορεί σήμερα η Ελλάδα να έχει αρχίσει να ανακάμπτει και να έχει ανάπτυξη και να μειώνει την ανεργία και να υπεραποδίδει στους συμφωνημένους δημοσιονομικούς στόχους έτσι ώστε να μπορεί η κυβέρνηση να δίνει και κοινωνικό πλεόνασμα για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά. Αλλά τα προβλήματα και τα ελλείμματα παραμένουν. Και το ερώτημά μου είναι προς το Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο που το ευχαριστώ για τη δουλειά του και δεν το καταγγέλλω τι θα κάνετε για να προασπίσετε τις ελεγκτικές σας δραστηριότητες απέναντι στην Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα που αρνείται να σας δώσει τα στοιχεία. Και προς την Κομισιόν, τι θα κάνετε εκτός από τσάι και συμπάθεια για να ενισχύσετε τη δημοκρατική λογοδοσία και τη διαφάνεια και να μην αποφασίζει για όλα πίσω από κλειστές πόρτες το Eurogroup. Και εσείς κυρία Πρόεδρε θα ενώσετε τη φωνή σας για να μπορέσει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να ζητήσει περισσότερη διαφάνεια και δημοκρατική λογοδοσία. κύριος Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Το Μάιο του 2016 κάνουμε μια ενδιαφέρουσα εκδήλωση μαζί με την κοινοβουλευτική ομάδα του ΑΛΔΕ και του S&D από την Ελλάδα με τίτλο «Λάθος μνημόνια, λάθος επιτροπή, λάθος κυβερνήσεις». Τώρα βλέπουμε 18 μήνες μετά την πολύ ενδιαφέρουσα και σημαντική και απόλυτα τεκμηρωμένη κριτική από το Ελεκτικό συνέδριο. Και λέμε 18 μήνες φαντάζεστε τι επίδραση είχαν στη ζωή των πολιτών και τι μας λένε για τα ευρωπαϊκά αντανακλαστικά. Σύμφωνα με τη σύσταση 3 του Ελεκτικού συνεδρίου, εάν η συνολική αναπτυξιακή στρατηγική μια χώρα δεν μπορεί να θεσπιστεί στο στάδιο έναρξη του προγράμματο, πρέπει να καθοριστεί όσο το δυνατόν συντομότερα. Η Ελλάδα στα πλαίσια του προγράμματος έκανε μια τεράστια δημοσιονομική προσαρμογή, που ακόμα όμως δεν ξέρουμε αν είναι βιώσιμη. Παράγει πρωτογενή πλεονάσματα από το 2013 και ταυτόχρονα παράγει και ύφεση, αδυνατή να αποκτήσει αναπτυξιακή δυναμική, παρότι η εφαρμογή των μνημονίων κρίνεται επιτυχής μέσω αλλεπάλληλων αξιολογήσεων εδώ και έξι χρόνια. Η Επιτροπή οφείλει άμεσα να αναπροσαρμόσει το πρόγραμμά τη και να λάβει μέτρα αναπτυξιακά. Ο στόχο για πρωτογενή πλεονάσματα 3,5% μέχρι το 2023 πρέπει να μειωθεί στο επίπεδο του 2% άμεσα. Το IMF αναγνώρισε τα λάθη των πρώτων προγραμμάτων και έχει αναπροσαρμοστεί. Η Επιτροπή πότε θα αναγνωρίσει τα δικά τη. Τώρα, στο τρίτο πρόγραμμα, επαναλαμβάνουμε τα ίδια λάθη. Και για να κλείσω. Ακούω από την κυβέρνηση και την Κομισιόν θετικού ρυθμού ανάπτυξη το 2017. Δεν είμαστε ευχαριστημένοι που η Ελλάδα μετά από 8 χρόνια ύφεση και σε ένα εξαιρετικά ευνοϊκό περιβάλλον παρουσιάζει ψήγματα ανάπτυξη. Και είναι θλιβερό η Επιτροπή να κρύβεται πίσω από αυτά τα ψήγματα αντί να χαράσει η ίδια τη στρατηγική ανάπτυξη αναλαμβάνοντα και τι ευθύνε τη. Πρέπει να ανοίξει αμέσω συζήτηση για το μνημόνιο 4 που δεν θα, είναι, δεν θα έχει δημοσιονομικού στόχου, έχει μόνο θεσμικού, με κύριο στόχο την ολοκλήρωση των διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων που χρειάζεται η χώρα μου όπω παραδείγματο χάρη τη βασικότερη οριζόντια μεταρρύθμιση τη δημόσια δίκη. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Σας ευχαριστώ. Ε, θα μιλήσω κι εγώ. Είμαι μέλος ε, και στην ομάδα για το πρόγραμμα για χρηματοπιστωτική βοήθεια στην Ελλάδα που παρακολουθεί, δεν θέλω να πω επιτηρεί την Κομισιόν να συνεισφέρω και εγώ κάποια πράγματα στην συζήτηση. Πρώτα απ' όλα τα προγράμματα βοήθεια της Ελλάδας είναι μια γιγάντια προσπάθεια αλληλεγγύης των Ευρωπαίων φορολογουμένων και αντιλαμβάνομαι βεβαίω ότι σώθηκαν και οι τράπεζες γιατί τις τράπεζες έχουν και οι απλοί άνθρωποι τους ε, λογαριασμούς τους. Πρόκειται για το κυκλοφοριακό σύστημα της ε, οικονομίας και βέβαια αφορά και τους αποταμιευτές ε, στην Ελλάδα και όλους. Και είδαμε ότι όταν η κατάσταση ε, κορυφώθηκε σε μια στιγμή επιβλήθηκαν έλεγχοι κίνησης κεφαλαίων και προσπαθήσαμε λοιπόν να κάνουμε κάτι και σε αυτό το μέτωπο. Να σας πω τώρα ότι αυτή η επίρρηψη των ευθυνών. Ακούω πολλά διάφορα, αλλά δεν άκουσα τίποτα για τις ευθύνες ε, της ε, ελληνικής κυβέρνησης και των ελληνικών κυβερνήσεων. Δηλαδή, ποιο είναι το αποτέλεσμα όταν εφαρμόζονται τα μέτρα μόνο εν μέρη. Και τα παλαιά λάθη βεβαίως είναι δραματικά και οποιοδήποτε άλλο κράτος θα το έφερναν σε αυτήν την ε, θέση. Και νομίζω ότι και το ύφος των παρατηρήσεων δεν συνάδει με την άνευ προηγουμένου αλληλεγγύη που έδειξαν ε, οι άλλες χώρες προς την Ελλάδα. Νομίζω ότι τελικά ο δρόμος ο οποίος ακολουθήθηκε αποδείχθηκε σωστός και πρόκειται για κάτι βεβαίως για το οποίο δεν είχαμε κάποια ε, εμπειρία και βεβαίως όταν ε, βγει η Ελλάδα εκτός ε, του ευρώ θα σήμαινε ότι σήμερα θα ήταν τελείως διαφορετική η συζήτηση που κάνουμε και η κατάσταση. Και βεβαίως κανείς δεν ξέρει και ποιες θα ήταν και για την Ευρωζώνη οι επιπτώσεις. Έρχομαι τώρα στο ελεγκτικό συνέδριο. με όλα αυτά τα οποία δεν ε, ήταν ε, γνωστά και όλα όσα έπρεπε να γίνουν πάρα πολύ γρήγορα από το 2009 και μετά ε, εγώ νομίζω ότι πολύ λίγα πράγματα πήγαν ε, στραβά. Πρόκειται δηλαδή για μια πάρα πολύ απότομη καμπύλη γρήγορης μάθησης. Βέβαια οπωσδήποτε μπορούν πάντα τα πράγματα να είναι καλύτερα. Αυτά και θα ήθελα τώρα να δώσω λόγο στην Κομισιόν για να απαντήσει. Σας ευχαριστώ. Θα ήθελα να επανέλθω σε δύο σημεία. Πρώτα απ' όλα για τα... τη θεσμική πτυχή. Αναφέρθηκε πολλές φορές, ε, η έκθεση αυτή αφορά μόνο την ε, Κομισιόν και θα ήθελα να υπενθυμίσω ότι όλα τα μνημόνια βασίστηκαν σε Κάποιου όρου στου οποίου συμφώνησαν όλα τα θεσμικά όργανα και το ΔΕΛΤΑΝΙΤΑΦ και σε συνεργασία με τι ελληνικέ αρχές. Μετά από μια μακροσκελή διαδικασία ιστορικών συζητήσεων και το ελεγκτικό συνέδριο επίση λέει σαφώ ότι αυτές οι διευθετήσει, αν και άτυπε ήταν αποτελεσματικέ. Αλλά επίση συνέστησε να επισημοποιηθούν, κάτι το οποίο δεχτήκαμε, και δώσαμε έμφαση στις ε, διαπραγματεύσεις ε, για να γίνει αυτό, αλλά αντιλαμβάνεστε ότι δεν μπορούμε εμείς να δεσμευτούμε για λογαριασμό άλλων που πρέπει να δεχτούν αυτές τις ε, διευθετήσεις ε, εργασίες που εξ ορισμού πρέπει να συμφωνηθούν από κοινού και επί της αρχής και επί της ουσίας. Τώρα, ρωτήσατε για το πρόγραμμα του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Σταθερότητας και εάν υπήρξαν κάποιες βελτιώσεις και από πολλέ ε, απόψεις είναι ένα βήμα προ τα εμπρό. Έχουμε ένα νέο νομικό πλαίσιο, μεγαλύτερη διαφάνεια και δημοκρατική λογοδοσία. Υπάρχει ενισχυμένο διάλογος με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και αυτό το οποίο είναι σημαντικό είναι η συνάφεια ε, η οποία ενισχύθηκε μεταξύ των στόχων της Ένωσης ε, και του μνημονίου. Πολύ μεγαλύτερη έμφαση δίνεται στην κοινωνική συνοχή και την απασχόληση και αυτό νομίζω είναι σημαντικό να το τονίσουμε. Τώρα, πού βρισκόμαστε αυτή τη στιγμή. Αυτή τη στιγμή που μιλάμε, σήμερα, έχει ξεκινήσει η τρίτη αξιολόγηση και βεβαίως ο συνάδελφός μου, ο επικεφαλής, είναι βεβαίως στην Ελλάδα, εκεί όπου πρέπει να είναι. Ελπίζουμε λοιπόν να ολοκληρωθεί σύντομα αυτή η αξιολόγηση και αναμένουμε το πρόγραμμα να τελειώσει κάποια στιγμή το επόμενο έτος και μετά θα δούμε το τι θα ακολουθήσει. Θα ήθελα επίσης να σας πω, επειδή το αναφέρατε κυρία Πρόεδρε, την ε, ομάδα εργασίας για την ε, οικονομική βοήθεια, όπως συμφωνήθηκε θα συνεχίσουμε εκεί τις επαφές μας, ε, θα συνεχίσουμε να ερχόμαστε να ενημερώνουμε το Κοινοβούλιο για την τρέχουσα κατάσταση. Ο συναδελφός μου, επικεφαλής της αποστολής, είναι ε, στην διάθεσή σας για να έρθει ε, βεβαίως και να σας ενημερώσει να πάει στιγμή. Ευχαριστώ. Κύριος Μουγκουρούσα, παρακαλώ. Σας ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Θα ήθελα εν συντομία να σχολιάσω κάποια από τα ζητήματα που ανέκυψαν. Καταρχήν για το Eurogroup. Όπως λέμε και στην έκθεση για τη σχέση μεταξύ Ευρωπαϊκής Επιτροπής και Eurogroup. Ούτως ή άλλως το Eurogroup είναι εκτός της εμβέλειας του δικού μας ελέγχου. Δεν μπορούμε να ελέγξουμε το Eurogroup και το αναφέρουμε στην έκθεση και αναφέρουμε ότι δεν ελέγξαμε ούτε τις πολιτικές αποφάσεις. Γιατί ούτε την απόφαση για την χορήγηση βοήθεια στην Ελλάδα, ούτε ε, δεν εξετάσαμε τι θα γινόταν στην Ελλάδα αν δεν είχε χορηγηθεί η συνδρομή, αν δεν εφαρμοζόταν πρόγραμμα και αν χρεοκοπούσε η χώρα δεν ελέγχουμε πολιτικούς ηθήνοντες. Δεν έχουμε τέτοια ελεκτική εντολή. Επίσης, δεν ελέγξαμε ούτε την ελληνική κυβέρνηση. Γιατί σε τελική ανάλυση η ελληνική κυβέρνηση έχει την ευθύνη της εφαρμογής των μέτρων που έχει υποσχεθεί να υλοποιήσει ως προαπαιτούμενα έγιναν κάποιες ερωτήσεις για τον προορισμό των κονδυλίων του προγράμματος. Τα προγράμματα δεν χρηματοδοτούν συγκεκριμένα σχέδια, αλλά συμπληρώνουν τις ε, ε, χρηματοπιστωτικές και οικονομικές ικανότητες της ελληνικής κυβέρνησης. Από αυτήν την άποψη η γνώμη μας για το πώς ε, εξελίχθηκε ο υπολογισμός του χρηματοδοτικού κενού των προγραμμάτων, δηλαδή τις ε, οικονομικές ανάγκες, χρηματοδοτικές ανάγκες της ελληνικής κυβέρνησης. Ε, για παράδειγμα, μία από αυτές ήταν η ανακεφαλαιοποίηση των τραπεζών. Και μία πολύ σημαντική ερώτηση που έγινε προς το ελεκτικό συνέδριο αφορούσε την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα. Όπως σας είπα και προηγουμένως, έχουμε δύο εκθέσεις ε, στις οποίες ε, μέχρι στιγμής ε, αντιμετωπίσαμε δυσκολίες για να ολοκληρώσουμε τον έλεγχό μας ως προς την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα. Δύο είδη ζητημάτων ανακύπτουν, προκειμένου. Από τη μία, Εμεί στο ελεκτικό συνέδριο έχουμε περιορισμένη εντολή, δηλαδή περιοριζόμαστε στην λειτουργική αποτελεσματικότητα μόνο της ΕΚΤ, γιατί αυτό προβλέπουν οι συνθήκες. Αυτή είναι η οριοθέτηση της εντολής μας. Και το δεύτερο αφορά την πρόσβαση στι πληροφορίε. Και για τα δύο αυτά θέματα έχουμε ξεκινήσει κάποιο προβληματισμό και θέλουμε να βελτιώσουμε τις σχέσεις μας με την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, να βρούμε ένα πρωτόκολλο συνεννόησης. Επίσης, εσείς ε, στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, ε, οι πολιτικοί θύνοντες δηλαδή και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, που είναι η αρμόδια για την νομοθετική πρωτοβουλία, μπορεί να ε, σχεδιάσει, να ενισχύσει, να αναπροσδιορίσει την εντολή μας απέναντι στην ΕΚΤ και εμείς το Ελεκτικό Συνέδριο, ως Ευρωπαϊκό Θεσμικό Όργανο, δεν έχει μόνο την ισχύ και το δικαίωμα ελέγχου, αλλά και το καθήκον ελέγχου. Θα μπορούσαμε να εξετάσουμε και τη θέσπιση άλλων μέτρων. Προς το παρόν όμως δεν έχει ληφθεί καμία απόφαση σχετικά. Πάντως όντως το θέμα μας προβληματίζει, μας απασχολεί και θα συνεχίσουμε τις εργασίες σχετικά. Ευχαριστώ. Και τέλος. Ε, Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ξέρω ότι θέλετε να τελειώσουμε τη συνεδρίασή μας στις 3.30, αν και το θέμα αυτό είναι εξαιρετικά ενδιαφέρον και περίπλοκο και θα Έπρεπε να το συζητήσουμε πιο εις βάθος σε περίπτωση που έχουμε να αντιμετωπίσουμε παρόμοια κατάσταση στο μέλλον. Η μεγάλη, το μεγάλο ερωτηματικό είναι η στόχοι δεν υλοποιήθηκαν όλοι. Η πραγματική οικονομική ανάπτυξη και βιώσιμη ανάπτυξη ε, θέλαμε. Θα πρέπει λοιπόν να σκεφτούμε γιατί δεν επετεύχθη αυτός ο στόχος. Θα, θα, θα έπρεπε βέβαια και η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα να ήταν πιο συνεργάσιμη. Τα όσα ακούσαμε σήμερα ε, να πω ότι ήταν πολύ θετικά η δουλειά του ηλεκτρικού συνεδρίου επίσης και θα συνεχίσουμε να συζητάμε το θέμα. Σας ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ. Θα πάει η Επιτροπή μας και στην Ελλάδα. Θα ευσκεφθούμε πάνω από 100 έργα προτεραιότητας, ε, έχουμε πάνω από 100 έργα προτεραιότητας, ε, επισκεφθούμε κάποια για να δούμε και την εκτελεσή τους, παραδείγματος χάρη αυτά τα οποία χρηματοδοτούνται από το Ταμείο Μετανάστευση. Σας ευχαριστώ για τη συζήτηση. Τελείωσε η συνεδρίαση και ακολουθεί αμέσως η συνδιαλλαγή. Σας ευχαριστώ.